Συνάδελφοι, επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι δήλωση της Επιτροπής για το κράτος δικαίου στην Ρουμανία. Δίνω το λόγο πρώτα πρώτα στην κυρία Γιούροβα για να μιλήσει εξ ονόματος της Επιτροπής. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, η Κομισιόν ξεκαθάρισε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και παραπέρα, ότι παρακολουθεί εκ του συνεγγύς και με πολύ μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις που αφορούν το κράτος δικαίου στη Ρουμανία. Ε, επανειλημμένα έχουμε πει ότι η Ρουμανία θα πρέπει να επιστρέψει στην μεταρρυθμιστική διαδικασία και μάλιστα κατεπηγόντως. Αυτό σημαίνει να πάει προς τα μπρος, όχι προς τα πίσω και να απόσχει από οποιοδήποτε βήμα που ε, ουσιαστικά αναιρεί την πρόοδο των προηγούμενων ετών. Η Κομισιόν και συγκεκριμένα ο πρώτος αντιπρόεδρος, ο Φρανς Τίμερμανς, προσωπικά έχει δεσμευτεί με την Πρωθυπουργό Νταντσίλα και οι εμπειρογνώμονε συναντήθηκαν πολλές φορές για επικοδομητική συζήτηση και διάλογο. Η Κομισιόν πάντοτε ξεκαθάρισε ότι <laughs> ο διάλογος για χάρη του διαλόγου δεν θα αρκεί και ε, αναμένουμε συγκεκριμένε δράσεις από την ρουμανική πλευρά και μάλιστα πολύ σύντομα. Η Επιτροπή συζήτησε την κατάσταση πριν δύο εβδομάδες. Δυστυχώς δεν ε, μπορέσαμε ακόμη να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι έχει επανέλθει στην ορθή οδό η Ρουμανία. Αν ε, δεν ε, διασκεδαστούν οι ανησυχίε μα, θα πρέπει να αναλάβει δράση η Κομισιόν και να χρησιμοποιήσει τα μέσα που έχει στη διάθεσή τη. Η σημερινή συζήτηση δεν αφορά τεχνικά ζητήματα ή να σα ενημερώσω ε, για ε, την ε, υπαναχώρηση που είδαμε στι συστάσει του μηχανισμού CVM. Εκεί υπάρχει τελμάτωση. Ή να συζητήσουμε ότι οι τελευταίε εξελίξει νομοθετικέ στη Ρουμανία για τη μεταφορά πολλών οδηγιών στο εσωτερικό δικαίωμα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανησυχίε με πιθανή συμβατότητα με το ευρωπαϊκό δίκαιο ή να αναφέρουμε περαιτέρω διάβρωση ε, της ε, εμπιστοσύνης και διάφορες ε, αυθαίρετες διαδικασίες διορισμών. Ε, επίσης, η διαδικασία για την επιλογή της ε, μελλοντική Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ε, δεν έχει συνεισφέρει στην επίλυση του προβλήματος. Βλέπουμε επαναχώρηση στο κράτος δικαίου στη Ρουμανία και κυρίως σε ό,τι αφορά την αμεροληψία του δικαστικού σώματος και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Καταρχήν, οι πιθανέ τροποποίησει ε, του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινική δικονομία. Ε, τέτοια θεμελιώδη ζητήματα χρειάζονται πολύ προσεκτική προετοιμασία, ε, διαβούλευση με το δικαστικό κλάδο και τα ενδιαφερόμενα μέρη και πολύ σαφή κατανόηση των αλλαγών. Οποιοδήποτε δράση αναλυφθεί θα πρέπει να συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς υποχρεώσεις καθώς και με τις συστάσεις του μηχανισμού CVM, όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς οι ρουμανικές αρχές ε, θα ε, αναλάβουν κίνδυνο αν προχωρήσουν ε, χωρίς να ακολουθήσουν μια τέτοια διαδικασία και αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να έχουμε μια de συστημική ατιμωρησία για υψηλούς αξιωματικούς που έχουν καταδικαστεί για διαφθορά. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το ανώτατο κυρωτικό δικαστήριο ε, και μία πιθανή συνέχιση μίας ε, δικαστικής απόφασης ε, που ζήτησε στον αλλάξη σύνθεση πέντε δικαστικών σχηματισμών δεν ε, μπορούμε να διαχωρίσουμε αυτό το θέμα από τις σημαντικές ε, συνέπειες του να ξανανοίξουν παλιές υποθέσεις. Ε, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζική παρέμβαση στην αμεροληψία της δικαιοσύνης. Ο κίνδυνος μαζικού προβλημάτων στο ρουμανικό ποινικό σύστημα και πάρα πολλών περιπτώσεων διαφθοράς δεν μπορεί να γνωριθεί. Τρίτον, το θέμα των διορισμών των εισαγγελέων και συγκεκριμένα η ανάγκη για ένα εύρωστο και αμερόληπτο σύστημα του διορισμού των επικεφαλής εισαγγελέων. Αυτό δεν είναι ένα νέο θέμα, όμως ο μηχανισμός ελέγχου και ισορροπιών έχει καταψηφιστεί. Επιτυχώς το αποτέλεσμα είναι μία επίμαχη διαδικασία για το να διεριστούν οι ενότατοι εισαγγελεί. Ο Γενικός Εισαγγελέας ε, και ε, ο επικεφαλής εισαγγελέας ε, καταπολέμησης διαφθοράς. Επίσης, ε, τα τμήματα ε, της εισαγγελία ε, που έχουν να κάνουν με το διορισμό των ανακριτών. Έχουν αναφερθεί ανησυχίες στην έκθεση CVM από την Επιτροπή της Βενετίας και από τον Γκρέκο. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση ενισχύει τη δομή αυτή. Όλα τα στοιχεία αυτά, όλα τους, προκαλούν μεγάλες ανησυχίες ε, αν τα δούμε και μεμονωμένα. Ενώ όλα μαζί ουσιαστικά δημιουργούν μια ιδιαίτερα ανησυχητικόνα. Τους τελευταίους μήνες ε, είδαμε μια ιδιαίτερα σταθή κατάσταση στη Ρουμανία με μια σειρά βιασμένων αποφάσεων ε, που ελήφθησαν και ουσιαστικά ζητήματα. Αν οι ανησυχίε αυτέ δεν διασκεδαστούν, η Κομισιόν θα πρέπει να δράσει και να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή τη. Επομένως, η Κομισιόν παροτρύνει τη Ρουμανία να ε, διαβουλευθεί και να φτάσει σε μία συνένεση, να ακολουθήσει τις συμβουλές της Επιτροπής της Βενετίας, ε, καθώς και τις διαδικασίες του CVM. Δεν είναι πολύ αργά για τη Ρουμανία για να ε, επανέλθει στις μεταρρυθμίσεις. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρέσλε, δύο λεπτά για το ΕΛΚ, έχει το λόγο. Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, δυστυχώ δεν μπορούμε να καλωσορίσουμε και την Προεδρία παρά το γεγονό ότι θα ήταν ε, πάρα πολύ ε, καλή να, παρα, να παραστεί εδώ η Προεδρία. Θα πρέπει να σα πω ότι ανησυχώ, ανησυχώ, γιατί ποτέ δεν έχουμε τόσο γρήγορα δει κατάρρευση του κράτου δικαίου όπω στη Ρουμανία και αυτό δεν έχει παρουσιαστεί σε κανένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω η Ρουμανία να αποτελέσουν την εξαίρεση. Και καλό θα ήταν να είχαμε ε, δράσει και να έχει δράσει η Ρουμανία πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο άμεσα. Αυτό που έχουμε να προτείνουμε προτείνουμε βάσει του άρθρου 7 να σταματήσουν οι πόροι, γιατί δεν μπορούμε να προστατεύσουμε του πόρου αυτού δεδομένη και τη κατάρρευση του κράτου δικαίου, γιατί η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για την είναι από ό,τι φαίνεται υπερβολικά επιβαρημένη η Προεδρία ή η ρουμανικη κυβέρνηση είναι και θύμα και θήτης. Και το πρώτο θύμα είναι η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, γιατί ουσιαστικά προωθείται έτσι η διαφθορά. βλέπουμε λοιπόν έναν πρόεδρο α, της, από τους σοσιαλιστές του Κοινοβουλίου, ο οποίος α, κατηγορείται και α, η, αυτή η ιστορία θα πρέπει να ακολουθηθεί και από του σοσιαλιστές και δημοκράτες γιατί αυτά τα δύο μέτρα και σταθμά είναι κάτι πολύ αρνητικό. Και βλέπουμε λοιπόν α, ε, α, ε, τη διαδικασία της ε, εισαγγελέως, της πρώην εισαγγελέως, η οποία κατηγορείται με διάφορα προσχήματα διαρκώς για εκδίκηση. Είναι υποψήφια των δύο μα, μεγάλων κομμάτων για τη νέα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα για να προστατευτεί η εισαγγελέας, υποψήφια εισαγγελέας και υπάρχει διάθεση να ανταμείψουμε ακόμα για την Ρουμανία για την παρτυπή αυτή. Αυτό πραγματικά δεν πρέπει να το αφήσουμε να συμβεί γιατί η Η υποψηφία του ταυτή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί μεν οικεί σε ό,τι αφορά κατάφορε παραβιάσει του κράτου δικαίου. Κυρίε και κύριοι, το θέμα λοιπόν είναι όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το θέμα είναι η αξιοπιστία και τη Επιτροπή του πρώτη του Αντιπροέδρου και όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρο. Και έχουμε μία μπλε κάρτα, κυρία Κρέσλε. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε την μπλε κάρτα. Θα ρωτήσω λοιπόν την εξή ερώτηση στα αγγλικά και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Τερμενία. Είπατε στην παρέμβασή σας ε, κάποια τρομερά πράγματα για το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ρουμανίας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πώς μπορείτε να εξηγήσετε στους Ρουμάνους ότι στη δική σας χώρα τα μέλη του συνταγματικού δικτύου μπορούν να είναι και κομματικά στελέχη, μέλη του κόμματος. Σας ευχαριστώ. Αγαπητέ συνάδελφε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή. Δεν είπα ότι το συνταγματικό Δικαστήριο έχει πολιτικά κίνητρα. Το θέμα είναι αν οι πολιτικοί ε, τηρούν το δίκαιο εγώ προασπίστηκα τι αποφάσει του συνταγματικού δικαστηρίου για την υποποίηση από του πολιτικού. Αυτό είναι το θέμα. Και έχει έρθει το πρόβλημα του χρόνου οι σοσιαλιστέ να, να τοποθετηθούν από αυτόν. Γιατί να ψηφίσουν λοιπόν οι Ρουμάνοι όταν πρόκειται για ρουμανικά ζητήματα. Αυτό είναι θέμα ολόκληρη τη Ευρώπη. Εγώ το είδα και στην υποψήφια του Εθνικού Συνεδρίου δεν μας είπε την αλήθεια τουλάχιστον. Το λιγότερο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που είχε. Το είδαμε για του υποψηφίου, την υποψήφια για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πότε επιτέλους ε, οι σοσιαλιστές θα αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά σαν ευρωπαϊκά θέματα. Δεν είναι ρουμάνικο το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Συντό συγγνώμη, λέει η πρόεδρο. Συνεχίζεται η συζήτηση. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο Ιωζεφ Βάιντεν Χόλτσερ από του Σοσιαλιστέ. Ευχαριστώ πολύ. Αντίθετα με αυτά που είπε η προελαλήσασα, πιστεύω ότι η Ρουμανική Προεδρία η οποία έχει πετύχει πάρα πολλά στο σύντομο χρονικό διάστημα που είχε στη διαθέσή τη. Πολλά κατάφερε λοιπόν να πετύχει παρά τις αντίξωε συνθήκε. Γι' αυτό λοιπόν, μα κύριε Πρέντα, ακούστε με, σας παρακαλώ λίγο ε, πειθαρχία. Γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο περίεργο το γεγονός ότι σήμερα αυτή η κατεπίγουσα συζήτηση πρέπει να γίνει. Αυτό το θέμα δεν το συζητάμε για, σε πρώτη φορά. Για πρώτη φορά, το Νοέμβριο το Κοινοβούλιο ξεκαθάρισε σε ψήφισμα ότι το θέμα της δικαιοσύνης και των ποινικών διώξεων στην ε, Ρουμανία δεν ε, μπορεί να απειλεί την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος αν θέλουμε να καταπολεμούμε την διαφθορά. Ο έλεγχος και ο έλεγχος θα πρέπει να εγγυώνται και ο κοινοβουλευτικό έλεγχος ε, των ε, μυστικών υπηρεσιών. Δυστυχώ, ε, οι αξιώσει μα δεν ε, λήφθησαν σοβαρά υπόψη. Αυτό μα λυπεί ιδιαίτερω. Το θέμα λοιπόν δεν είναι συγκεκριμένα να στραφούμε κατά τη Ρουμανία. Το θέμα είναι η κοινή ερμηνεία του δικαίου. Ένα εύρυθμα λειτουργών κράτο αποτελεί πυλώνα τη κοινή Ευρώπη. Και αυτό σαφώς θα ορίζεται στα κριτήρια της Χάγης. Η τήρηση λοιπόν των κριτηρίων αυτών και η αιμονή στην τήρηση των κριτηρίων δεν αποτελεί θέμα ιστορικό ενό κράτου μέλου. αποτελεί ε, κάτι που αφορά όλους μας και φυσικά δεν μπορεί να γίνεται μονομερός και να αποφασίζεται μονομερός, αλλά τα κοινά αυτά, οι κοινέ αυτές αρχές θα πρέπει να καθορίζονται μέσω διαλόγου. Αυτό είναι το μήνυμα που έχουμε να στείλουμε προ το Βουκουρέστι. Μόνο έτσι θα μπορέσει να αναπτυχθεί από κοινού η Ανατολή και η Δύση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρο, Και τώρα το λόγο έχει η Μόνικα Μακοβέη από το ECR. Σήμερα στη Ρουμανία μια ομάδα διαφθαρμένων πολιτικών ε, με επικεφαλή στον καταδικαστέντα Ντράγκνε, ο οποίος τελεσίδικα έχει καταδικαστεί και έχει και νέες δίκες, ε, κρατάει όμοιρο ε, τη χώρα, δεν ε, σέβεται το πρόγραμμα διακυβέρνηση που είχαν ανακοινώσει στις εκλογές, αλλάζουν το νόμο, σβήνουν παραβιάσεις και ουσιαστικά πολιτικά ασκούν έλεγχο στους δικαστές και χρησιμοποιούν χρήματα από τις επενδύσεις για να δίνουν μίζες, καταστρέφουν την έννοια της δημοκρατίας προκειμένου αυτή η οι πολιτικοί να την κλειτώσουν από τη δικαιοσύνη ε, και ε, τελικά κρατούν ε, όμερους 20 εκατομμύρια ανθρώπους για να σωθεί μόνο ένας. Οι Ρουμάνοι δεν είναι αδρανείς. Εδώ και δύο χρόνια βγαίνουμε στο δρόμο. μας ρίχνουν δακρυγόνα, μας χτυπάνε, μας ρίχνουν πλαστικές σφαίρες ή χειροβομβίδες. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να κατεβαίνουμε στο δρόμο. Και Στη συνέχεια ο δρόμος μας είναι η Ευρώπη. Βλέπουμε με απελπισία την καταβήθηση της χώρας ε, που ε, τη χτυπούν ο Ντράγνε, ο Ταριτσάνου και άλλοι. Εγώ όμως δεν μπορώ να σιωπάσω, δεν μπορώ να ε, μας κρατούν όμοιροι κάποιοι εκατοντάδες πολιτικοί που ασκούν την εξουσία σας. Ζητώ να βοηθήσετε την Ρουμανία, γιατί η Ρουμανία σήμερα ζει μια εγκληματική δικτατορία και την τραγωδία του αδιάσματος της χώρας. 4 εκατομμύρια Ρουμάνοι έχουν φύγει μόνο τα τελευταία χρόνια. Η απομάκρυνσή μας από την Ευρώπη είναι ο εφιάλτης που ζήσαμε εδώ και δεκαετίες. Αυτό είναι το τελευταίο τρένο το οποίο μπορούμε να πάρουμε. Θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Έντφελντ, για τρία λεπτά. Yes, thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ την Επίτροπο. Ξεκινώ λέγοντας ότι συμφωνώ με την ενόχληση της κυρίας Γκρέσλε για την απουσία του Συμβουλίου. Πόσο μάλλον που η Προεδρία είναι η χώρα την οποία συζητούμε. Μη χειροκροτάτε ακόμα. Μπορεί να μην σας αρέσει αυτό που θα πω μετά. Λυπάμαι επίσης διότι δεν είναι εδώ ο κύριος Τίμερμανς. Δεν θέλω να σας προσβάλλω κύριε Επίτροπε, αλλά είναι ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για το θέμα. Τι έκανε για το θέμα αυτό τα τελευταία πέντε χρόνια. Την περασμένη εβδομάδα μόνο υπέβαλε η Επιτροπή μία ανακοίνωση για το κράτος δικαίου που στην ουσία δεν άξιζε το χαρτί που ήταν πάνω στο οποίο ήταν ε, γραμμένη. Και δεν εμφανίστηκε καν ο κύριος Τίμερμαν στην Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών για να το παρουσιάσει. Πού είναι σήμερα, ε, τι έκανε τελευταία πέντε χρόνια. Εγώ πραγματικά κουράστηκα να συζητώ σήμερα για την Ρουμανία, λείπει το ΕΛΚΑ. Αύριο Ουγγαρία, οι σοσιαλιστές θα κριτικάρουν, θα επικρίνουν τους... Ε, το, το, το, το ΕΛΚ. Ξέρω ότι κάποιοι φωνάζουν γι' αυτό, δεν θέλω να το πω όλου. Ε, η κυρία Γκρέσλε διαμαρτύρεται, αλλά το θέμα γίνεται τελικά πάντα κομματικό. Δεν είναι κομματικό το θέμα. Το θέμα είναι για τις αξίες που περιλαμβάνει το άρθρο 2 της συνθήκης που μας αφορούν όλους ανεξάρτητα από το πολιτικό μας χρώμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δυόμιση χρόνια πριν το Κοινοβούλιο υιοθέτησε μία θέση, μία, υπέβαλε μία πρόταση για ένα γενικό μηχανισμό κράτους δικαίου που καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη, όλες τις κυβερνήσεις. Η Επιτροπή και δεν με έμφωμα εσά, κύριε Επίτροπε, ο κύριος Τίμερμαν είναι ο υπεύθυνο. είπε δεν το χρειαζόμαστε γιατί έχουμε όλα τα εργαλεία στην εργαλειοθήκη που χρειαζόμαστε. Δεν τα έχουμε. Ο κύριος Τίμερμαν είναι candidate και ο κύριος Βέμπερ το ίδιο. Υποψήφιοι για πρόεδρο της Επιτροπής και οι δύο. Γιατί λείπουν και οι δύο υποψήφιοι? Τι προτίθεται να κάνουν όταν, αν γίνουν πρόεδροι της Επιτροπής. Ο πρόεδρος της Επιτροπής κύριος Βέμπερ θα κάνει αυτό που υπερψήφισε ως ευρωβουλευτής. Δηλαδή θα προτείνει πλήρη μηχανισμό προστασίας του κράτους δικαίου που θα αφορά όλα τα κράτη-μέλη. Τελειώνω, πρόεδρε. Η ομάδα μου, η φιλελεύθερη, σαφώς και ξεκάθαρα απομακρύνθηκε από το αδελφό Ρουμανικό κόμμα. Όχι μόνο για παραβιάσεις ε, ε, ε του Ευρωπαϊκού Κράτους Δικαίου, αλλά για μια σειρά άλλων νομοθετικών κειμένων ε, ε, γάμο για όλους. Ε, είμαστε εξαιρετικά απογοητευμένοι από τη συμπεριφορά και την προσπάθειά τους να εμποδίζουν την ε, καταχώρηση και τις υποψηφιότητες νέων, ευρω... νέων κομμάτων που θέλουν να κατέβουν στις ευρωεκλογέ. Ευχαριστώ. Υπάρχει μια μπλε κάρτα κύριε Πρέντα. Συμφωνώ με την επίκρισή σας για την επιτροπή και τον κύριο Τίμερμανς, κύριε Ιντενβέλτ και δεν θέλω να κάνω κομματική συζήτηση, αλλά ο κύριος Φερχόφστατ, επικεφαλής της ομάδας σας, δεν είπε τίποτα μέχρι. Σιώπησε. Ε, το πρόβλημα δεν ξεκίνησε πριν από τρεις μήνες. Όταν είχαμε ζητήσει να κάνετε κάτι, μείνατε ε, στο περιθώριο. Τώρα μετράτε την, την κατάσταση εν ώψη των εκλογών και εσείς κυρία μου. Γιατί ο κύριος Φεχόφστατ, πείτε μου, δεν είπε τίποτα τότε από πολιτική φιλία ε, με τον κύριο Τριτσάνο, από, μετράνε περισσότερο οι προσωπικές φιλίες από την πραγματικότητα, πείτε το μου. Λάθος κάνετε. Δείτε τα πρακτικά της Ολομέλειας. Η στάση της ομάδας μας ήταν πάντα ξεκάθαρη. Αν ήταν εξίσου ξεκάθαρη και η θέση του ΕΛΚ, δεν θα είμαστε στην κατάσταση που είμαστε τώρα με την Ουγγαρία. Είμαστε εξαιρετικά αρνητικοί και κριτικοί σε αυτά που συμβαίνουν στη Ρουμανία. Επίσημα απομακρυνθήκαμε από το κόμμα των φιλελευθέρων που είναι στην συγκυβέρνηση σαν Ευρωπαϊκό Κόμμα και ζητήσαμε την απομάκρυνσή τους από την πολιτική μας οικογένεια. Το κάνουμε με βαριά καρδιά διότι έχουμε πολλά χρόνια πολιτικής φιλίας όντως, αλλά εμείς τιμούμε τις αρχές μας αντίθετα από το ΕΛΚ που ακόμα και τώρα δεν απομακρυνθήκε πλήρω από τον κύριο Όλμπαν. Διαβάστε λοιπόν τα πρακτικά της Ολομέλειας. Εγώ προσωπικά κύριε Πρέντα είχα συμμετάσχει στις συζητήσεις για τη Ρουμανία και ήμουν εξαιρετικά επικριτική. Να είστε κι εσείς εξίσου σε ό,τι φέρω το δικό σας μέλος, τον κύριο Όρμπαν. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σελτζαντίνη. Ο... Ε, έχετε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Μποστινάρο και στην κυρία Ενετφέλτ. Δέχεστε. Μουλτσομέσκ. δέχεστε. ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι συνάδελφε, δύο σύντομες ερωτήσεις για σας. Ξέρετε πόσες φορές ε, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ρουμανίας χαρακτήρισε τις πράξεις τη κυρία ε, Κεβίση ε, ω αντισυνταγματικέ. Ξέρετε πόσες φορές διαπιστώθηκε ότι παραβίαζε το Ρουμανικό Σύνταγμα και μετά έχουμε την υπόθεση που γνωρίζετε τις κατηγορίες περί κατάχρησης αξιώματος. Οι σημαντικότερες μαρτυρίες προέρχονται από δύο εισαγγελείς της Εθνικής Διευθύνσης Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Αυτοί μαρτυρούν κατά αυτής, είναι οι βασικοί μάρτυρες. Πώς μπορείτε λοιπόν να μιλάτε για πολιτική πίεση σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για δικαστικών υποθέσεων, αλλά πόσο ξέρω πρόσφατα το δικαστήριο αποφάσισε ότι η κυρία Κεβίση, μπορεί να τελειώσω. Θέλετε να με ακούσετε. Σας ενδιαφέρει η απάντηση. Έχω 30 δευτερόλεπτα και τα μισά πέρασαν ήδη. Αυτό που ξέρω είναι ότι πρώτα απ' όλα το δικαστήριο ήδη επέτρεψε στην κυρία Κιόβεση να ταξιδέψει και να εκφραστεί. Το θέμα είναι ότι τα επιχειρήματα που ακούω πάντα είναι... δεν κάνουν τα πράγματα καλύτερα, διότι η εικόνα που έχουμε εδώ είναι ότι υπάρχει ένα απόλυτο χάο. Και χρειαζόμαστε ένα κράτο δικαίου, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για το ρουμανικό λαό, διότι οι νέοι άνθρωποι στη Ρουμανία διψούν για μια χώρα σταθερή, ε, για μια κυβέρνηση αξιόπιστη, μη διεφθαρμένη. Και ακούμε όλες τις ιστορίες, ε, ένα στο δικαστήριο, ε, οι μυστικές υπηρεσίες που παρεμβαίνουν. Όλα αυτά κάνουν τα πράγματα καλύτερα, δεν νομίζω. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε τη συζήτηση κυρίας Αρτζεντίνα από τους Πράσινους. Δεν, ε, το κράτος δικαίου δεν είναι αριστερό ή δεξιό και είναι πολύ οδυνηρό που βλέπουμε ότι η ρουμανική κυβέρνηση στηρίζει την Ουγγρική μην βάζοντας στην ημερήσια διάταξη την έκθεση για την Ουγγαρία. Όλοι το είπαν, αλλά είναι πολύ απογοητευτικό. Η Ρουμανική Προεδρία δεν είναι εδώ. Απίστευτα πράγματα. Επίσης, ε, η Προεδρία απονομιμοποιεί τον υποψήφιο του Κοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και έτσι απονομιμοποιεί όλη τη διαδικασία. Η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι κρίσιμη στο κράτος δικαίου. Και έχουμε μια χώρα η οποία συνεχώς υπαναχωρεί και προεδρεύει και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τούτη την ώρα. Άλλο παράδειγμα. Ξέρω τον Ιανουάριο του 2011 όταν η Ουγγρική κυβέρνηση είχε την προεδρία του Συμβουλίου Πάλι ένα εξάμεινο δεν έγινε τίποτε. Πραγματικά πρέπει να ντρέπονται γι' αυτό. Έξι εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογέ και έχουμε αυτή την κατάσταση εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλώ ήρθατε αγαπητοί συνάδελφοι. Εκ μέρου του ΙΕΝΕΦ, ο κ. Μπάτεν. Ο κ. Μπάτεν δεν είναι εδώ. Περνάμε στον κύριο Λενάρ για ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση χωρών που έχει συμπράξει για να δώσει έναν, μια μάχη ε, και να συνενώσει δυνάμεις. Αυτό γίνεται πάνω στη βάση ισχυρών θεμελίων κοινών αξιών μόνο. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση σήμερα. Και είδαμε έλλειμμα στις αντιδράσεις της Κομισιόν και η Πολωνία επίσης πρέπει να υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 7. Έχουμε και τη Ρουμανία, έχουμε τη Μάλτα που δεν τις έχουμε προσέξει ε, ιδιαίτερα, αλλά πρέπει να εστιάσουμε στη Βαλέτα και τον Βουκουρέστι. Δεν πρέπει να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μπορούμε να προβάλλουμε την ένωσή μας, να τη στηρίξουμε όταν τα μέτρα είναι τα ίδια για όλους. Δεν πρέπει να παίζει ρόλο ε, η φιλία με το δικαστήριο στην περίπτωση της Μάλτας και της Ρουμανίας θα πρέπει άπαξ και διαπαντός να υπάρξει παρέμβαση της Κομισιόν. Ο κύριος Νίκα, ε, λεπτά. Ξαναγίνεται μια συζήτηση προεκλογική. Είναι μια συζήτηση για την οποία πρέπει να πούμε πως ε, τελικά δεν μιλάμε για την Ρουμανία. Πολύ συχνά λέμε πράγματα χωρίς να είμαστε σαφής. Ποια είναι η κατάσταση του κράτους δικαίου. Χωρίς ελευθερίες για τους πολίτες δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Το 2009 στη Ρουμανία υπογράφηκε ένα μυστικό πρωτόκολλο με την ε, μυστική υπηρεσία πληροφοριών. Αυτό το μυστικό πρωτόκολλο βγήκε στο φως, διέρευσε και αυτό αποκάλυψε σημαντικές παρανομίες και καταχρήσεις. Η Ρουμανία λοιπόν έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά στη δικαιοσύνη της. Σε οτιδήποτε έχει σχέση με τα δικαιώματα των πολιτών. Τα ρουμανικά φαρμακευτικά προϊόντα, για παράδειγμα, δεν, έχουν τις, ε, δεν τυχαίνουν τις ίδιες με, μεταχείρισης με άλλα προϊόντα της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Το ίδιο και στα αεροδρόμια ε, στου λιμένε. Από τη μια μεριά πηγαίνουν Ρουμάνοι, από αλλού πηγαίνουν οι υπόλοιποι. Ε, το 90% των Ρουμάν πολιτών θεωρεί ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν ε, θεωρούν ε, καλέσει τι παραβάσει και τι καταχρήσει που έχουν γίνει στη δικαιοσύνη. Στη Ρουμανία ο πληθυσμός, η κοινή γνώμη είναι πολύ ευαίσθητη σε θέματα δικαιωμάτων λόγω του κομμουνιστικού παρελθόντος. Δεν θέλουμε να εκβιαζόμαστε. Δεν θέλουμε να ε, κινηματογραφείται η προσωπική ζωή των εισαγγελέων στην Ρουμανία προκειμένου να εκβιαστούν μετά. Θέλουμε να μας μεταχειρίζονται με, τους ίδιους, ε, με τον ίδιο τρόπο ε, που μεταχειρίζονται τους πολίτες σε όλες οι υπόλοιπες χώρες. Αυτοί που έχουν αυτιά ας ακούσουν και αυτοί που έχουν μάτια ας δουν. Η Ρουμανία ε, αξίζει περισσότερο. Ευχαριστώ. Η κυρία Βέμπερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η Ρουμανία έχει ενταχθεί στο μηχανισμό αξιολόγηση και ε, του του κράτους δικαίου ε, της Κομισιόν και έχει επικριθεί για πρακτικές ε, σχετικά με την απόδοση δικαιοσύνης. Πριν από μερικές εβδομάδες, ε, αρχηγοί ε, κρατών κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν από τα δικαστήρια της Ρουμανίας να σταματήσουν έρευνα που γίνεται εναντίον ε, γίνονται σχετικά με Ρουμάνο πολίτη ε, που είχε υποστεί παραβίαση των δικαιωμάτων του. Το Ανώτατο ε, Δικαστικό Συμβούλιο της ε, Ρουμανίας είπε ότι ο Ταγιάννη, ο Φερχόφστατ και ο Βέμπερ μέσω των δηλώσεών τους θέτουν πίεση στους εθνικούς δικαστές που έχουν αναλάβει αυτή την υπόθεση και υποσκάπτουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στη Ρουμανία. Οπότε, συνάδελφοι, θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αρχίστε να συμπεριφέρεστε Όπω ζητάτε από τους άλλου πολιτικούς να συμπεριφέρονται. Ευχαριστώ. Ο κ. Πρέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λυπάμαι που δεν εκπροσωπείται εδώ η ρουμανική κυβέρνηση, <laughs> παρόλο ότι το θέμα μας είναι ακριβώς η Ρουμανία. Κανείς δεν εκπροσωπεί εδώ λοιπόν την Προεδρία του Συμβουλίου. Αυτό δείχνει την περιφρόνηση που δείχνει το Συμβούλιο προς το όργανό μας. Είναι πραγματικά κρίμα σε αυτή την πρώτη Ρουμανική Προεδρία να βρισκόμαστε σε τέτοια κατάσταση. Κάποιος θα έπρεπε να είναι εδώ. Όμως το καθεστώς του Βουκουρεστίου ε, δεν συνδέεται πλέον με το κράτος δικαίου. Η πλειοψηφία που κυβερνά τη χώρα από το 2016 κάνει αυτό που είπε ο κ. Νίκα. <laughs> Ε, πιέζει τους εισαγγελείς και τους δικαστές και δημιουργεί ε, θεσμούς που θα οδηγήσουν, θα επιτρέψουν στην αναθεώρηση τελεσίδικων αποφάσεων ε, αποφάσεις που είχαν ληφθεί προκειμένου ε, να καταπολεμηθεί η ε, διαφθορά. Ο πρόεδρος τους έχει καταδικαστεί δύο φορές για διαφθορά, αυτός ο αστείος τύπος. Δείξτε μου μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, κυβερνάται από τέτοιο άνθρωπο. Άνθρωπος ο οποίος παρέμεινε στο αξίωμά του έχοντας καταδικαστεί δις. Καταδικάστηκε για απάτη. Πώς είναι δυνατόν να δεχόμαστε συμμαχίες τέτοιων ε, ανθρώπων που θα καταστρέψουν τη χώρα μας. Ευχαριστώ. Κυρία Γκραπίνη. Και κυρία Γκραπίνη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ ε, αγαπητοί συνάδελφοι, να κάνω μια παρατήρηση. Αυτή η συζήτηση είναι μια αποτυχία, κυρία Επιτροπή. Το βλέπετε και από τον κόσμο που είναι εδώ. Δύο άνθρωποι είναι εδώ. Οι σημαντικότεροι ηγέτε δεν είναι εδώ, είναι δειλοί. Ε, θα έρθετε στη Ρουμανία, στη χώρα μου κύριε Βέμπερ και θα πείτε ε, να σταματήσει μια υπόθεση ενώπιον των δικαστηρίων. Κύριε Επίτροπε, ξέρετε ότι στον τομέα της δικαιοσύνης δεν μπορείτε να πάτε σε μια κυβέρνηση και να τους πείτε τι θα κάνουν. Ακόμη και αν είστε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και οι παρεμβάσει ε, των Ευρωπαίων αξιωματούχων έχουν επηρεάσει αρνητικά τη δικαιοσύνη στη Ρουμανία. Οι πολίτε στη Ρουμανία δεν καταλαβαίνουν γιατί ορισμένοι αξιωματούχοι και ευρωβουλευτέ ε, θέλουν να παρέμβουν σε υποθέσει ενώπιον ρουμανικών δικαστηρίων. Ναι, ε, είμαστε σε προεκλογική φάση. Ναι, το καταλαβαίνω, ναι. Ο κύριο Πρέντα το είπε ότι και εσεί έχετε προεκλογική εκστρατεία αυτή τη στιγμή. Οπότε το ΕΛΚ προσπαθεί αυτή τη στιγμή να κερδίσει κάτι από αυτή την εκστρατεία. Ε, Επίτροπε, θέλω να πείτε στου Ρουμάνου ότι δεν δώσατε ούτε ένα παράδειγμα παραβίασης του κράτου δικαίου, ούτε ένα. Η ρουμανική κυβέρνηση έχει μια επιτυχή προεδρία. Λυπάστε που είχαν τόση επιτυχία, που ολοκλήρωσαν τόσα θέματα και τόσα αρχεία. Γιατί το κάνετε αυτό. Πέρυσι είχαμε ένα ψήφισμα, ήταν άδικο και το ξέρετε. Ξέρετε ότι υπάρχει κάτι σε αυτό το ψήφισμα το οποίο δεν θα λέγατε για καμιά άλλη χώρα. Ε, κατηγορείται τη Ρουμανία που άλλαξε τον επικεφαλής ε, ενός φορέα, ε, ο οποίο κατέστρεψε το φορέα αυτό, τη δικαιοσύνη. Μιλάμε για τις ζωέ χιλιάδων ανθρώπων, χιλιάδε δίκε που ακόμη και εσείς είχατε πει ότι έπρεπε να ξαναγίνουν. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους ε, να υποφέρουν από την αδικία. Ποιον προστατεύεται η Ρουμανία. Δεν είναι ε, ένας άνθρωπος, ε, είναι 20 εκατομμύρια άνθρωποι. Ο κύριος Πρέντα παρακαλώ. Θα δώσω τον κύριο, λόγο στον κύριο Χεκμάρκ. Κυρία Πρόεδρε, το να υπονομεύουμε την ανεξαρτησία του δικαστικού, η υπονόμευση Τη ανεξαρτησία των εισαγγελέων, η παρεμπόδιση τη δημιουργίας νέων κομμάτων, απόπειρα νομιμοποίηση τη διαφθορά, καταπολέμηση όχι της διαφθορά, αλλά αυτών που καταπολεμούν τη διαφθορά, το να σε ενοχλητικούς ηγέτε ανεξαρτήτων φορέων, απαγόρευση εξόδου τους από τη χώρα, Φυσικά και μιλάμε εδώ για μια κατάρρευση του κράτους δικαίου. Και αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι η άρνηση. Αλλά πρέπει να πω όμως, ε, ε, κύριε Βιντεχόζερ, ότι η σιωπή των σοσιαλιστών είναι εκοφαντική. Η συμβολή σας εδώ, απόψε, δεν ήταν εντυπωσιακή, αλλά και θα σας πω γιατί η υπεράσπιση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας δεν ακολουθεί κομματικές γραμμές. Η κατάχρηση της εξουσίας στην Ουγγαρία και στην Πολωνία δεν αιτιολογεί την κατάχρηση εξουσίας στη Ρουμανία και άκουσα πολλούς από εσάς να το λέτε ε, πολύ ηχηρά για την Ουγγαρία όπως και εγώ και για την Πολωνία. Αλλά η σιωπή σας είναι εκοφαντική. Καταχράστε τη υποχρέωσή σα να υπερασπίζεστε τη δημοκρατία. Εσεί, ω ηγέτε, εδώ απόψε τη ε, ομάδα των Σοσιαλιστών, είστε λάθο. Το λόγο έχει ο κύριο Αρβαμά για ένα λεπτό και μισό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μα πού είναι ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς. Δεν βλέπω. Η Ρουμανική Προεδρία που είναι. Ούτε εκείνους τους βλέπω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε για να προωθήσει την ειρήνη, τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου. Όπως και οι άλλοι συνάδελφοι του ΕΛΚ, ανησυχώ πολύ για τη Ρουμανία και το κράτος δικαίου εκεί, δεδομένων των πρόσφατων εξελίξεων. Η Ρουμανία επιχειρεί να προχωρήσει σε αλλαγή του ποινικού κώδικα, ναι, αποποινικοποιώντας όμως τα διάκατη διαφθορά. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τις συνεχείς παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη ε, τα ειδικά τμήματα για τις έρευνες που ασκούν πιέσεις στους δικαστές και στους εισαγγελείς. Όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν. Ε, πρέπει η ρουμανική κυβέρνηση να σταματήσει να υποσκάπτει τις βασικές αξίες της Ένωσης. Αυτό πρέπει να είναι κορυφαία προτεραιότητα όλων μας. Επίσης, ε, κυρία Ίνφελ, θα σας συμβούλευα να δείτε καλύτερα την απόφαση του ΕΛΚ στις 20 Μαρτίου από το 20 Μαρτίου στις Βρυξέλλες. Νομίζω ότι δεν ανταποκρίνονται οι παρατηρήσεις σας στην αλήθεια αυτής της δήλωσης. Κύριε Μποστινάρο, περιμένετε. Μου ζητήσατε διαδικαστικό. Θα είναι μόνο αυτό, όχι άλλο σχόλιο. Ε? Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σας υπενθυμίσω κάποια πράγματα, αγαπητοί συνάδελφοι του ΕΛΚ ίσως δεν ήσασταν παρόντες αλλά η απόφαση του Συμβουλίου να μην εκπροσωπείται εδώ είναι απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων. Ζητήστε από τους αρχηγούς των ομάδων σας ε, πώς λήφθηκε αυτή η απόφαση. Θα έπρεπε να αναφέρετε ένα άρθρο. Ε. Δεν ε, κάνετε αναφορά στον κανονισμό. Κύριε Μωρίσα, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι, η Ρουμανία είναι φιλοευρωπαϊκή χώρα. Ο ρουμανικός λαός έχει ασπαστεί τις ευρωπαϊκές αξίες, την ειρήνη, την ελευθερία, το κράτος δικαίου, την προηγούμενη διετία εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους υπέρ των ευρωπαϊκών αξιών. Οι πολιτικοί έχουν υποχρέωση να ακούσουν τη φωνή του λαού. Οι πολιτικοί δεν επιτρέπεται να αλλάζουν τον νόμο προς ίδιων συμφέρον. Το ξαναλέω, εκατομμύρια... Ε, ε, Ρουμάνοι δεν θέλουν αμνηστία, δεν θέλουν συγχώρεση όλων αυτών. Θα πρέπει λοιπόν η ρουμανική κυβέρνηση να προχωρήσει στις αποφάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ρουμανική κυβέρνηση πρέπει να ακούσει τι λέει ο λαός. Ο πρόεδρος Ιωάννης στις 22 Μαΐου αποφάσισε δημοψήφισμα που θα δώσει την ευκαιρία στους Ρουμάνους να εκφράσουν την επιθυμία τους σε σχέση με το δικαστικό σύστημα. Μπορεί να πούνε όχι στην άφεση, στην αμνηστία, Μπορεί να πούνε όχι ε, στις ε, ε, αρνητικές τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα, ο οποίος πρέπει να αλλάξει λαμβάνοντας υπόψη την άποψη των δικαστών, των ειρηνοδικών και των εταίρων. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον ρουμανικό λαό στη μάχη που δίνει για τη δικαιοσύνη και τις ευρωπαϊκές αξίες. Μπλε κάρτα από την κυρία Γκραπίν, τη δέχεστε. Μάλιστα. Αγαπητέ συνάδελφε, έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Είπατε ότι άλλαξαν εν μια νυχτή νόμι; Ποιοι νόμοι? Εκτός από αυτόν που ανέφερε ο κ. Τσόλος. Ξέρετε κάποιο άλλο νόμο που να άλλαξε? Ευχαριστώ κυρία Γκραπίνη. Υπάρχει μια μακρά σειρά διαταγμάτων τα οποία έχουν εκδοθεί τον τελευταίο καιρό από αρχή, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2017, το 2013, την επόμενη μέρα εκατοντάδες χιλιάδες άτομα βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν. Τελειώσατε? Ωραία. Περνάμε στη διαδικασία του Catch the Eye. Κύριε Γιαροκά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θέλω να μιλήσω εναντίον των δύο μέτρων και δύο σταθμών. Ε, οι ίδιες κατηγορίες έχουν απευθεί και εναντίον της Ουγγαρίας. Παρ' όλα αυτά, η Ρουμανία έχει κάνει σημαντικότατη πρόοδο ό,τι αφορά την ένταξη των πιο φτωχών τμήματων του πληθυσμού. Ε, αντιθέτως, τα ε, ευρωπαϊκά κονδύλια φτάνουν πολύ καθυστερημένα και γι' αυτό το λόγο ε, θα πρέπει να συνεννοηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των Επιτρόπων και κυρία Κρέτσου, έτσι ώστε να φτάνουν χρήματα από τα διαχρονικά ταμεία έτσι ώστε να βοηθηθούν αυτοί οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν λαμβάνουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια αυτή τη στιγμή διότι υπάρχουν ε, γραφειοκρατικά προβλήματα. Και αυτό το λόγο ε, ε, διώκονται από τις αιστείες τους. Κριστέα η Επίτροπος κύριε Επίτροπε ε, είναι το δικό μας σχέδιο είναι ένα ευρωπαϊκό όραμα ο λαϊκισμός και οι ακραίες τοποθετήσεις ε, που αμφισβητούν το ευρωπαϊκό όραμα ε, έχουν ε, τις ρίζες τους στην πραγματικότητα του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μακριά από τους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, λάμπει δια της απουσίας της. Όταν βλέπουμε το τι έχει γίνει. Ε, απ' την άλλη μεριά σε άλλα θέματα ε, παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις ε, της χώρας. Δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρεμβαίνει στις δικαστικές και συνταγματικές υποθέσεις χωρών. Ε, μας χρησιμοποιείτε ως ε, πιόνι για να κερδίσετε κάποιους πόντους στις ευρωεκλογές. Το κάτσουδιά είναι ε, ομιλίες ενός λεπτού. Παρακαλώ πολύ να το σεβαστείτε. Ο λόγος στον κύριο Γιούρεκ. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι, κυρία Επίτροπε. Υπόθηκε ότι αν η κατάσταση στη Ρουμανία δεν αλλάξει, τότε η Κομισιόν θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Ευτυχώ η Επιτροπή αυτή δεν πρόκειται να λάβει πλέον κανένα μέτρο. Αρκετά μέτρα είδαμε από την Ευρωπαϊκή αυτή Επιτροπή. Μόνο εκλογικές κινήσεις μπορεί να κάνει τώρα Ρωτήσαμε γιατί δεν ήταν εδώ ο κύριος Τίμερμαντς. Πιστεύω ότι έχει συνηθίσει με εκλογικές κινήσεις τέτοιου είδους. Όσον αφορά τη Ρουμανία, η κατάσταση στη Ρουμανία είναι δύσκολη και περίπλοκη. Ε, το ίδιο όπως και στον Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν καταλαβαίνω τι ανοχή έχει η κυβέρνηση και στη μικρή διαφθορά, γιατί η διαφθορά είναι ένα γενικευμένο κακό. Αλλά αυτό που δεν μου αρέσει επίσης είναι η εποπτεία των πολιτικών και των πολιτών. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια πράγματα. Είναι πρόβλημα, αλλά οι Ρουμάνοι πρέπει να το λύσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Νικολάη, η σειρά Κυρία Πρόεδρε, η συζήτηση αυτή για το κράτος δικαίου, βασικό θεσμό της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν προκαλείται μια τέτοια συζήτηση και δεν ε, παρίσταστε εδώ, είναι, είτε είναι ότι περιφρονείτε τη συζήτηση ή περιφρονείτε τους πολιτικούς που συμμετέχουν στη συζήτηση αυτή. Δεν είναι σωστή αυτή η συζήτηση και φιλότιμη ε, μας προσβάλλει εδώ σε αυτό το ημικύκλιο, μας προσβάλλει από αυτούς που δεν συμμετέχουν. Έχει κανείς την εντύπωση ότι παίζει σε μια ταινία με κάποιον που καταδικάζεται για αυτά που σκέφτεται. Αυτό που θα κάνατε, αν είχατε ε, ένα ελάχιστο αξιοπρέπεια, ε, θα πηγαίνετε να δείτε τι έχει γίνει στη Ρουμανία. Δεν έχουμε υιοθετήσει καμία νομοθεσία και όμω μα επικρίνουν γι' αυτό. Αντιλαμβάνομαι πόσο σημαντικό είναι να μαζέψετε ψήφου ε, όσοι θέλουν να μείνουν στην εξουσία, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι αυτού του είδου συμπεριφορά απομακρύνει του πολίτε από την Ευρώπη. Πιστεύω ότι θα πρέπει να παρατήσετε το λαϊκισμό που βλέπουμε σήμερα. Ολοκληρώθηκαν εδώ. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα το Κατζιάι. Όλοι θα μιλήσετε, κυρία Βαΐ. Ευχαριστώ πολύ. Για να απαντήσω στην Επίτροπο Γιούροβα, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ξέρετε τον Ισφαν Μπέκε και έναν άλλον Ρουμάνο ε, που αντιμετωπίζει ποινική δίωξη. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα. Η πολιτική ασκεί πιέσεις στην ποινική δικαιοσύνη και ξαναζούμε ε, τις ε, πιο δύσκολες εποχές του, του όπου τους αντιπάλους, ε, οι πολιτικοί τους αντιμετώπιζαν με φυλάκιση και με ποινικέ διώξεις για να επιτύχουν τους πολιτικούς τους στόχους. Έχουμε δύο πολίτες ε, εδώ που αντιμετωπίζουν ποινικέ διώξεις ενώ το μόνο που έκαναν ήταν να δώσουν μάχη για τα ε, δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας στη Ρουμανία. Τα γνωρίζετε αυτά. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ο κύριος Πόπα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε. Και πάλι δεν πρόκειται για συζήτηση, πρόκειται για μια φιέστα προεκλογική όπως άλλωστε ήταν και ο σκοπός αυτών που άρχισαν τη συζήτηση. Δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο, δεν υπάρχει ουσία. Δεν θέλουμε να μπούμε σε ε, ουσιαστικές λεπτομέρειες. Κανείς δεν θέλει να γίνει συγκεκριμένος. Μιλάμε γενικά για φόβους, ανησυχίες, κινδύνους. Κυρία Επίτροπε, πρέπει να ανησυχούμε, πρέπει να μιλάμε για κινδύνους όταν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Στρασβούργο υπαγορεύουν στους ε, Ρουμάνους δικαστές τι πρέπει να κάνουν. Αυτό είναι απαράδεκτο. Το κράτος δικαίου σημαίνει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Δεν επιτρέπεται να υπαγορεύεται όποιοι κι αν είστε ε, τι θα, στη δικαιοσύνη τι θα κάνει. Κυρία Ταπεντέν. Κυρία, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Θα αρχίσω με μία ερώτηση. Μιλάμε για το κράτος δικαίου. Εννοούμε βέβαια και σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών. Γιατί αυτό θέλουμε να κάνουμε στη Ρουμανία. Θέλουμε ένα σύστημα δικαιοσύνης που θα είναι δίκαιο, που θα σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών, όπου δεν θα υπάρχουν καταχρήσεις από τους εισαγγελείς, ε, η ζωή και η σταδιοδρομία των ανθρώπων δεν θα καταστρέφονται. Το μήνυμα μου προς όλους τους ε, βουλευτές ε, που χρησιμοποιούν σλόγγαν τη Ρουμανία στην προεκλογική τους εκστρατεία είναι «Έχετε εκλεγεί γιατί είστε αξιόπιστοι τα μάτια των ψηφοφόρων. Δεν επιτρέπεται τώρα να γίνει μια συζήτηση ακόμη η οποία ε, επιτίθεται σε ένα κράτος μέλος. Αυτό ε, εισάγει διπλά μέτρα και δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εδώ θέλετε να αποκομίσετε ωφέλη, αλλά αυτό υποσκάπτει το κύρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος ε, Τζάκον. Ευχαριστώ. Είναι δύσκολο να καταλάβω πώς μπορούμε να μιλάμε για ένα θέμα, το κράτος δικαίου, όταν αυτό δεν ορίζεται συγκεκριμένα. Στο βαθμό που η ποινική δικαιοσύνη αποτελεί εθνική αρμοδιότητα και υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των δικαστικών συστημάτων των κρατών μελών, δεν είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε ε, μια απόφαση. Γι' αυτό απλώς θορυβούμε θορυβούμε εδώ μέσα και τίποτε περισσότερο. Πρόκειται για μια εθνική αρμοδιότητα της Ρουμανίας και βεβαίως το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ρουμανική Δικαιοσύνη θα λειτουργεί με βάση τις ευρωπαϊκές αξίες και τους κανόνες, αλλά ε, πέραν αυτού πρέπει να πω ότι δυστυχώς δεν έχουμε κράτος δικαίου, ε, χρειάζεται πολλή δουλειά για να φτάσουμε εκεί. Περιμένω όμως από το επόμενο κοινοβούλιο να ορίσει το κράτος δικαίου και να το θέσει σε εφαρμογή. Κυρία Πρόεδρε, συναδελφοί, κυρία Επίτροπε, η ε, Ρουμανία είναι η χώρα μου και ποτέ δεν θα επιτρέψω να κυκλοφορούν ψεύδι ε, σε βάρος της. Υπάρχει κράτος δικαίου στη Ρουμανία. Το λέω και το τονίζω. Κάποια ρουμανικά πολιτικά κόμματα προσπαθούν να παρουσιάσουν στον ε, δημόσιο χώρο μια τελείως διαφορετική εικόνα. Για αυτό ωφελεί την αντιπολίτευση, κάποια ευρωπαϊκά κόμματα και γι' αυτό ε, ε, διαστρεβλώνεται τελείως η εικόνα της ε, δικαιοσύνης στη Ρουμανία. Εκείνοι που κατηγορούν είναι οι ίδιοι που ασκούν πιέσεις στη δικαιοσύνη στην χώρα μου προσπαθώντας να επιβάλλουν καταδίκες, ποινές, ακόμα και λήψη αποδεικτικών στοιχείων και ασκούν πιέσεις στους δικαστές για να αθωώσουν κάποιους δικούς τους. Όταν τα μέλη της ρουμανικής αντιπολίτευσης εντοπίσει κάποια αμφιλεγόμενα θέματα από, από νομικής άποψης ε, σταματούν ε, να σκουν πιέσεις. Αυτό που βλέπετε σήμερα διακοπή. Εγώ ήμουν υπέρ της ε, ένταξης της Ρουμανίας ε, δεν ήθελα να μείνει στην άκρη η Ρουμανία και να υπάρχει δικαιοστάσιο. Ήμουν ε, μεταξύ εκείνων που ε, καταπολέμησα τη διαφθορά, την εκμετάλλευση των παιδιών. Μετά από 15 χρόνια βλέπω ότι η Ρουμανία ασκεί την Προεδρία, δεν ε, μπήκε στον κόπο να έρθει εδώ και έχει δημιουργήσει ε, ε, ε, εγκληματική οργάνωση η οποία αποσπά ενωσιακά κονδύλια. Θα πρέπει να μην διστάσουμε να καταγγείλουμε αυτά που γίνονται στη Ρουμανία. Όπως είπε και η Επίτροπος Γιούροβα, πρόκειται για το κράτος δικαίου στην Ένωση, όχι μόνο στην Ρουμανία εδώ. Θέλουμε να στηρίξουμε τους ε, ε, ε, αθώους Ρουμάνους πολίτες που αψήφισαν κινδύνους κρύο για να διαδηλώσουν υπέρ του κράτους δικαίου. Ο κ. κυρία κύριε Επίτροπε, ως σοσιαλιστής παρεμβαίνω. δεν μιλώ ούτε στα ουγγρικά ούτε στα ρουμανικά ε, σε, σεβόμενος την παρουσία αυτών των χωρών. Ε, ο, η συζήτηση για το κράτος δικαίου πολύ συχνά καταλήγει να γίνεται ε, διαξυφισμός κατηγοριών. Ε, στο άρθρο, από το άρθρο, στο άρθρο 7 εντάχθηκαν διάφορες χώρες όπως γνωρίζετε και δεν θέλω αυτές οι χώρες ε, να ανταλλάσσουν κατηγορίες με τις υπόλοιπες. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το βασικό είναι ότι έχουμε πολλά να κάνουμε μπροστά μας. Ε, χρειαζόμαστε ένα αξιόπιστο μηχανισμό επαλήθευσης ε, του κατά πόσον πληρούνται οι αρχές του άρθρου 12 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κράτος δικαίου, θεμελιώδη δικαιώματα, ποιότητα της δημοκρατίας και καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτός ο μηχανισμός, κυρία Γιουρόβα, είναι κάτι το οποίο απαιτούμε εδώ και καιρό από την Κομισιόν, εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Κομισιόν θα πρέπει στην επόμενη θητεία να υποβάλει προτάσεις για ένα τέτοιο μηχανισμό. Ευχαριστώ. Ο λόγος στην κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, να εκφράσω την πεποίθηση ότι εκπροσωπώ όλη την Κομισιόν, το σύνολο του οργάνου. Αυτό για όσους επικρίνουν την απουσία του κυρίου Τίμερμανς, του πρώτου αντιπρόεδρου. Ο κύριος Τίμερμανς ε, προσπαθεί εντατικά να διατηρήσει ανοιχτό τον πολιτικό διάλογο με τη ρουμανική κυβέρνηση και είναι ο τελευταίος ο οποίος θα πρέπει να επικριθεί ε, για οτιδήποτε έχει κάνει για οποιαδήποτε παράληψή του. Δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω είναι το εξή. Η Κομισιόν δεν παρεμβαίνει σε συγκεκριμένε δικαστικές υποθέσεις. Αυτό το αναφέρω προς την κυρία Γκραπίνη. Αυτή είναι η αρχή μας. Δεν παρεμβαίνουμε. Εξετάζουμε μόνο συστημικά προβλήματα που προκύπτουν από την ομοθεσία της χώρας. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε αναφερθεί στις πρόσφατες ε, ε, μεταρρυθμίσεις που έγιναν στο δικαστικό σύστημα στη Ρουμανία. Γιατί το συνολικό αθρηστικό αποτέλεσμα όλων αυτών των αργών μπορεί να οδηγήσει σε παράβαση του κράτους δικαίου στη Ρουμανία. Τελευταίο μου σχόλιο. Κυρία Μοργκάη, όχι, δεν γνωρίζω αυτές τις δύο περιπτώσεις, Μπέκε και Σουίτς. Θυμάμαι μου στη δική μου περίπτωση, τη δική μου υπόθεση από το 2006. Εγώ κατηγορήθηκα για διαφθορά το 2006. Στο πλαίσιο μιας πολύ βρώμικης υπόθεσης ε, που έγινε μοναδικό γνώμονα πολιτικά συμφέροντα και αμαυρώθηκε η εικόνα μου στα μέσα ενημέρωσης και θυμάμαι τον εαυτό μου. Ούτε για ένα δευτερόλεπτο δεν πίστευα ότι, δεν πίστεψα ότι κάποιος δικαστής θα με έστελνε στη φυλακή πίστευα στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη στη χώρα μου. Και επί τη ευκαιρία να σας πω ότι η υπόθεση δεν έφτασε καν στα δικαστήρια ποτέ. Ήτανε απλώς λάσπη. Το θυμάμαι πολύ καλά όμως. Και είναι παράδοξο το ότι η Ρουμανία μου προσέφερε δουλειά μετά από αυτό. Γιατί όλα είχαν καταστραφεί, όλη μου η καριέρα μέχρι η οικογένειά μου είχε καταστραφεί. Δούλεψα στη Ρουμανία, η Ρουμανία μου έδωσε μια ευκαιρία να χρησιμοποιήσω τη γνώση μου, να την προσφέρω και γι' αυτό είμαι ο, ο τελευταίος άνθρωπος που θα πρέπει να κατηγορηθεί ότι φέρεται κατά της Ρουμανίας. Στην Ρουμανία μπορεί να φτάσουμε στην κατάθεση στάση σημεία αναστρέψιμων αλλαγών του δικαστικού συστήματος με συστημικές παραβάσεις του κράτους δικαίου της ε, ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας του δικαστικού συστήματος. Αυτοί, αυτές κινδυνεύουν. Πολύ στενά παρακολουθώ το τι κάνει η Ρουμανία μέσω του μηχανισμού CVM ε, και ανησυχώ για τις αλλαγές που ξεκίνησαν ξαφνικά προς λάθος κατεύθυνση ενώ όλα πήγαιναν προς τη σωστή κατεύθυνση πριν. Η, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι σημαντικός πυλώνας του δημοκρατικού καθεστώτος του δημοκρατικού συστήματος και έχει αναπτυχθεί εδώ και πολλές δεκαετίες σε όλα τα κράτη-μέλη είναι μια αργή προοδευτική διαδικασία που οδηγεί σε ένα ισορροπημένο συνταγματικό σύστημα. Ο δικαστικός πυλώνας είναι βασικό κομμάτι αυτού. Μπορεί όμως να καταστραφεί. Εν μια νυχτή, πραγματικά εν μια νυχτή. Και αυτό θέλει να αποφύγει η Κομισιό στη Ρουμανία. Οπότε ο διάλογος συνεχίζεται. Θα συμφωνήσω με αυτούς και αυτές που είπαν ότι οι Ρουμάνοι και οι Ρουμάνες αξίζουν περισσότερα, θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Οι συζητήσεις γίνονται σε τεχνικό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Θα ζητήσω να επιστρέψει σε πολιτικό επίπεδο ο διάλογος και να είναι θετικός, επικοδομητικός, να οδηγήσει σε θετικές αλλαγές και στην επάνωδο των μεταρρυθμίσεων στη σωστή άκουσα. Ευχαριστώ. Δεν σας δίνω το λόγο. Ήρθατε τελευταία στιγμή. Δεν ζητήσατε μπλε κάρτα. Δεν μπορείτε να θέσετε μπλε κάρτα για την κυρία Γιούροβα. Εάν λοιπόν δεν έχετε κάτι διαδικαστικό με κάποιον αριθμό και μην μιλάτε και σε, χωρίς μικρόφωνο, δεν έχει νόημα. Ζητώ συγγνώμη. Έπρεπε να είχατε έρθει λίγο νωρίτερα για να συμμετέχετε σε αυτή τη συζήτηση